Now, um, we would start by submitting... Uh, Θα αρχίσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μήπως υπάρχει κανένα σχόλιο υπ' Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα υπάρχει τίποτε για τα πρακτικά της 11ης και 12ης Ιανουαρίου. Όχι ε, τότε εγκρίνονται και αυτά. Και τώρα το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Κούκαν θα αρχίσει την παρουσίαση των συμπερασμάτων της αντιπροσωπείας του. Ορίστε κύριε Κούκαν μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συναδέλφοι. Στη 12η διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ ΕΚ και Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ιδίως συζήτησαν όλα τα προβλήματα της χώρας και η συζήτηση ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη μερικές φορές αλλά ειλικρινής. Ως προς την πρόοδο προς την ένταξη επανειλημμένως δηλώθηκε από μας ότι η χώρα έχει καθυστέρηση σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της περιφέρειας, της περιοχής εκείνης. Δύο εκθέσεις προόδου, το 8 και το 9, αναφέρουν ότι η πρόοδος είναι πολύ αργή για την πλήρωση των κριτηρίων σταθεροποίησης που προβλέπει η Συμφωνία Σύνδεσης. Αυτό το είπαμε επανειλημμένος και δεν φάνηκε κανένα ενθουσιασμός ως αντίδραση από τους άλλους. Επίσης συζητήσαμε την ανάγκη που υπάρχει για συνταγματική μεταρρύθμιση ώστε να υπάρξει ένα πιο συνεπές γενικό σύστημα δικαστικό και συνταγματικό θεσμικό γιατί χρειάζεται ανεξάρτητο κοινοβούλιο. Αυτό είναι σαφές. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις αναφέρθηκαν επίσης και ως προς την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δεκεμβρίου στις περιπτώσεις Σέντιτς και Κίντιτς, όπου λέει ότι το Σύνταγμα προβλέπει άνηση μεταχείριση των πολιτών που δεν ανήκουν στους τρεις ιδρυτικούς λαούς γιατί τους εμποδίζει να είναι υποψήφιοι στην Προεδρία ή στο Κοινοβούλιο. Η δε ημερομηνία για την πιθανή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ε, συζητιέται ακόμα από τους πολιτικούς εκεί. Ίσως χρειαστούν πολλές εβδομάδες ακόμη μέχρι να εγκριθεί η μεταρρύθμιση. Οι περισσότεροι βουλευτές ήταν μάλλον αρνητικοί και τόνιζαν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί λίγος ο χρόνος πριν τις εκλογές και τα λοιπά, οι οποίες προβλέπονται για τον Οκτώβριο. Εμείς τονίσαμε ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου. Για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ήταν θετικά τα αποτελέσματα και η Βοσνία Ριζεγοβίνη εκπλήρωσε όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η Κομισιόν προετοίμαζε την τρίτη της επίσκεψη εκεί. Οι δύο προηγούμενες είχαν θετικά αποτελέσματα. Τονίσαμε ότι εδώ είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι όταν οι πολιτικοί ενώνονται για να πετύχουν έναν κοινό στόχο όλα είναι δυνατά και ότι το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν και για άλλα θέματα. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους πολίτες της χώρας και ήταν το κύριο θέμα συζήτησης και με τους εκπροσώπους των Μίκη όμικρων οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς την χορήγηση του δικαιώματος αυτού πριν τις εκλογές λέγοντας ότι τα κόμματα θα κάνουν κατάχρηση για δικούς τους λόγους. Απ' την άλλη χαιρετήσαμε την συμφωνίες με την Κροατία και τη Σερβία για τις αμοιβέ εκδόσεις. Η εντυπωσιακή ανέχεια στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ευθύνεται εν μέρη, ε, οφείλεται εν μέρη και στην γενική κρίση αλλά και στην απουσία οικονομικών μεταρρυθμίσεων υπενθυμίσαμε στις αρχές ότι πρέπει να πληρώσουν όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Αμείου και είπαμε ότι πρέπει να κάνει και μια πραγματική και σωστή απογραφή για να έχουμε σωστά δεδομένα γιατί η έλλειψη στατιστικών στοιχείων θα βλάψει τη χώρα και ως προς τις ενταξιακές της προοπτικές και θα καταστήσει πιο δύσκολη την επίλυση σημαντικών κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων. Γενικά αποσαφηνίσαμε ότι η όλο και πιο εθνικιστική ρητορία που ακούγεται δημόσια στη Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές αξίες και καταδικάσαμε στεναρά οποιασδήποτε προσπάθειες αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και υποστηρίξαμε πλήρως την υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ που ζήτησε να εφαρμοστούν πλήρως οι αποφάσεις της. Σας είπα ότι στις αρχές του Οκτωβρίου θα γίνουν εκλογές και πρέπει τα πολιτικά κόμματα να φερθούν υπεύθυνα, να μην κάνουν κατάχρηση της ευκαιρίας αυτής για εκμετάλλευση εθνικιστικών αισθημάτων και στόχων και να μην λένε ότι δεν γίνεται, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα κλπ. Η αντιπροσωπεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης δεν συμφωνούσε ότι γενικά είναι αρνητική πολιτική κατάσταση, αν και αυτό φάνηκε και από την κοινή δήλωση όπου οι εκπρόσωποι του κόμματος του Ντόντιτς ήθελαν να διαγραφούν όλες οι αναφορές στην υπάτη αρμοστία. Γενικά κύριε Πρόεδρε όλες οι προσπάθειες μέχρι τώρα που έχουν γίνει για να προοδεύσει η χώρα απέτυχαν να επιφέρουν αποτελέσματα. Πρέπει όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει τον διάλογο ενεργά γνωρίζοντας ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξουν αποτελέσματα γρήγορα. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν, διασκέψεις, συναντήσεις κλπ. Για να ζητήσουμε από τους πολιτικούς τους, να πούμε στους πολιτικούς τους ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μεν το πολιτικό μέλλον της χώρας, αλλά ότι εκείνοι είναι υποχρεωμένοι να πετύχουν αποτελέσματα και να εφαρμόσουν τα κριτήρια. Η αντιπροσωπεία μας έδειξε μεγάλη ενότητα και αυτό το μήνυμα μετέφερε προς όλους. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πακ τώρα. Θα ήθελα να συμπληρώσω μόνο μερικά πράγματα. Η συνεδρίαση στο Σαράγεβο έδειξε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στα κεφάλια, στα μυαλά των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο. Κανένας δεν κάνει βήματα προς τον άλλον για μια νέα τάξη, για μια ενίσχυση του συνολικού κράτους της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Και πιστεύω ότι έχουμε πολύ δύσκολους καιρούς ακόμα μπροστά μας. Ούτε θα λυθούν τα θέματα αυτά με τις επόμενες εκλογές. Το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, αν θα γίνει πριν μετά τις εκλογές, είναι τελείως άσχετο γιατί δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα κόμματα. Και όλα αυτά τα κόμματα δεν θέλουν να κάνουν ούτε σπιθαμή, ούτε ρούπι δεν το κουνάνε προς τη κοινή συμβίωση. Ο καθένας προσπαθεί να περάσει τις δικές του απόψεις. Συνένεση, συμβιβασμός, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, όπως έχουμε γνωρίσει εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό ε, και είναι πολύ καλός πολιτής. Πουλάει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ούτε τους διευθυντές δεν διορίζει των διαφόρων οργανισμών για να λειτουργήσει το κράτος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην κυβέρνηση την ίδια. Ήρθε σε μένα εκείνο πριν από ένα χρόνο και λέει ότι μιλάτε η διεθνή κοινότητα μόνο με τους ηγέτες των κομμάτων και όχι με τον ίδιο. Μα ο ίδιος τι είναι το μακρύ χέρι του κόμματός του στην κυβέρνηση. Γιατί να πάμε να μιλήσουμε με αυτό, να μιλήσουμε με τον αρχηγό του κόμματος κατευθείαν. Όλοι εξαρτώνται από κάποιους που τους έχουν στείλει στις θέσεις και στα αξιώματα που κατέχουν. Πραγματικά, ξέρετε ότι ασχολούμαι ε, από το 91 με την περιοχή αυτή και πάω στο Σαράγεβο και έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Ας πούμε ότι έγινε μια καλή αρχή για τη θεώρηση των διαβατηρίων και ήλπισα ότι εντάξει αφού τα βρήκαν εκεί θα προχωρήσουν και σε άλλους τομείς. Ε, δεν έγινε αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ και θα πρέπει να πω ότι μετά από αυτές τις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί απέναντι στην κυβέρνηση αυτή, όποια βγει, και τα κόμματα και να πούμε ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση είναι εκ των όνουκ άνευ. Τώρα έχουμε αυτή την περίπτωση Φίντσι που είναι οι άνθρωποι αυτοί που δεν είναι ούτε Βόσνοι, ούτε Σέρβοι, ούτε Κροάτες, οι λεγόμενοι λοιποί, the others, ε, ξαφνικά εξαφανίζονται, ε, να, να βγει δηλαδή αυτή η διάταξη από το Σύνταγμα και να ονομαστούν διαφορετικά. Ε, αυτοί οι others, οι λοιποί, είναι ένας τέταρτος. Γιατί έχουν μοιράσει όλα τα πόστα στα τρία. Αν έρθουν και οι άλλοι, λοιπόν, οι λοιποί θα έχουν και τέταρτη θέση. Ε, ποιοι είναι αυτοί. Έχουμε χιλιάδες μεικτούς γάμους. Τα παιδιά δεν μπορούν να δηλώσουν τι είναι, ούτε θέλουν να δηλώσουν, εν πάση περιπτώσει, οι μετάδε. Ζουν στη Βοσνία Ζαγοβίνη και είναι πολίτε. Δεν είναι οι άλλοι, δεν είναι οι λοιποί, οι others. Ε, και θα παρακαλούσα και τη Λάδη ε, Άστον να καταλάβει και ο κύριος Φίλιπ ότι εδώ διακυβεύεται και ένα ε, τμήμα της δικής μας αξιοπιστίας εάν αποτύχουμε στη Βοσνία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and I'm sure that this uh, will... Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά θα εκτιμηθούν δεόντως από τους συναδέλφους και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η κυρία Μουνιές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμμετείχα κι εγώ στην αντιπροσωπή αυτή και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κούκαν ε, για την ε, ηγεσία του, για τον τρόπο με τον οποίο προείδρευσε σε μια πολιτικά περίπλοκη κατάσταση, γιατί είναι πολύ δύσκολη στη Βοσνία Ζεκοβίνη. Πραγματικά δεν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά πολιτικών κομμάτων να γίνει κάποια πρόοδο, εν πάση περιπτώσει, προ την οικοδόμηση ενό κράτου με βάση τις συμφωνίες του Ντέιτον που ήταν πολύ καλές για την ειρήνευση αλλά δεν είναι αρκετές για την εδραίωση ενός κράτους οι συμφωνίες του Ντέιτον. Το πρόβλημα υπάρχει και είναι το πρόβλημα της ανθεώρησης του συντάγματος. Δεν θα προλάβουν τώρα με τις εκλογές και θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με τις εκλογές που δεν μπόρεσαν συμμετάσχει το 6-7% ε, στις εκλογές. Γιατί δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα αυτοί οι άνθρωποι να συμμετέχουν πουθενά. Ούτε θέλουν τα πολιτικά κόμματα, ούτε θέλει το Κοινοβούλιο να τους συμπεριλάβει. Επίσης υπάρχει μια δραματική διάκριση και διαχωρισμό κοινωνία των πολιτών και κομμάτων. Ε, συναντηθήκαμε με ΜΚΟ που μα ζήτησαν να παραλύσουμε εμεί μέχρι μετά τι εκλογέ την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων. Είναι απορία άξιο γιατί το ζητάνε οι πολίτε, η κοινωνία των πολιτών, για να μην νομιμοποιήσουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δράση αυτής της κυβέρνησης και αυτού του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουν και κυρίως τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις της Βοσνίας της ίδιας που θα πρέπει να τους δοθεί μια όθηση, κάποια ενθάρρυνση να παροτριθούν, να έχουν κίνητρα, δεν ξέρω κάτι να κάνουν, να προχωρήσουν στη θεσμική μεταρρύθμιση, στην αθεώρηση του συντάγματος, στον πραγματικό εκδημοκρατισμό και οικοδόμηση ενός κράτους και να μην διαλύονται σε διάφορες ενότητες, οντότητες, κοινότητες και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αρχάς Φεβρουαρίου η ομάδα μας, ε, η Φιλελεύθερη, επέστειλε επίσης αντιπροσωπεία στη Βοσνία Ριζαγοβίνη και στο Σαράγεβο και στην Πάνια Λούκα. Και είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Και εγώ είμαι πεπισμένη ότι ήταν πολύ σημαντική η συμφωνία του Ντέιτον, καλή και άγια, το 1995 όμως. Ε, θα πρέπει τώρα να είμαστε πολύ ρεαλιστές, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να αναθεωρήσουμε τα πράγματα. Διότι η πολιτική ευθύνη στη χώρα δεν είναι στα χέρια των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αυτής. Αλλά στα χέρια της διεθνούς κοινότητας. Και αυτό ε, εμποδίζει να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτου προέλευσης τοποθέτηση. λένε ότι αν δεν υπάρχει η ευθύνη στα χέρια τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν. Τους βολεύει όμως, τους αρέσει να τρέχουν τα κόμματα στον ύπατο εκπρόσωπο και να κλαίγονται και να γκρινιάζουν και να με ψηρινούν, να παίρνει αυτές τις αποφάσεις για να μην τις παίρνουν οι ίδιοι. Αν θέλουμε λοιπόν να φέρουμε πιο κοντά τη Βοσνία Ζεγοβίνη στην Ευρώπη και να τη βοηθήσουμε στις ευρωπαϊκές τις προσδοκίες και προοπτικές, ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ύπατος εκπρόσωπος εκεί. Και ταυτόχρονα ε, βέβαια είναι και θέμα ασφαλείας αυτό. Στη χώρα είναι σοβαρό και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και ακούσαμε σε πολλές συνεδριάσεις ότι εκκρεμεί η κατάσταση αυτή, η ασφάλεια είναι αρκετά εύθραυστη ακόμα, εξού και η διεθνή στρατιωτική παρουσία θα πρέπει να παραμείνει. Ακόμα και όταν φύγει ο υπατός εκπρόσωπος. Και η κατάργηση της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης ένα αρνητικό αποτέλεσμα της συμφωνίας του Dayton. Η διεθνή κοινότητα και το Dayton έχτισαν και ένα σύστημα που ε, προώθησε τη διέρεση, τον διχασμό των πολιτών. Ορισμένοι δεν συμμετέχουν στην πολιτική ζωή γιατί δεν έχουν το δικαίωμα καν Ευτυχώ υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου του Στρασβούργου που την αντίθετη κατεύθυνση. Χρειάζεται χρόνο για τη συμφιλίωση. Και κάτι που μας ανησύχησε ιδιαίτερα στη δική μας αντιπροσωπεία ήταν ότι όταν ακούσαμε ότι οι νέοι στη χώρα, η νέα γενιά είναι επίσης πάρα πολύ διχασμένη. Πάνε σε διαφορετικά σχολεία, δεν συνεννοούν, δεν επικοινωνούν καν μεταξύ τους και μακροπρόθεσμα η προοπτική, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, με τη λεγόμενη βοήθεια εντός εισαγωγικών ε, του γραφείου του ΙΠΑ, του εκπροσώπου και της διεθνούς κοινότητας, είναι, πώς να το πω, δεν πρόκειται να προχωρήσει η χώρα, έχει αποτελματωθεί και μάλλον θα επιστοδρομήσει και σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των διαβατηρίων της θεώρησης. Είναι φυσικό τους δικαίωμα, λέει, και, θα πρέπει να, και το αξίζουν. Βέβαια πρέπει να ανταποκριθούν και εκείνοι τι υποχρεώσεις τους. Αλλά να απελευθερώσουμε τα διαβατήρια και τις θεωρίες τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And, uh... Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μποσκούρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ στα αγγλικά, κυρία Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν για την παρουσίασή του και να θέσω και ένα ερώτημα. Γιατί η κυρία Πάκα σε ότι η κατάσταση εκεί με τα πολιτικά κόμματα είναι δύσκολη. Όταν είχαμε συναντήσει τον κύριο Ρίνσκο είπε ότι Υπάρχει ένα καινούργιο κόμμα εκείνο του σκηνοθέτη που είχε πάρει το Όσκαρ που νομίζω έχει ως τίτλο «Το κόμμα μας» και ότι είχε την πρόθεση να φροντίσει τους πάντες και τους μικρούς γάμους και τα λοιπά, όχι εθνικιστικά δηλαδή. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Κούκαν, συναντήσατε τους εκπροσώπους και του νέου αυτού κόμματος Ευχαριστώ, κύριος Λούνατσεκ. Ε, ε, Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου ομάδα έχει έρθει η Μαρία Κορνέλισεν. Δυστυχώς σήμερα ακολύεται και απουσιάζει. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε αυτό που είπε και η κυρία Πακ και κάποια άλλη ήδη η κατάσταση είναι περισσότερο από προβληματική, ε, το θέμα του συντάγματος δηλαδή. Και δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω αυτό που ήδη υπόθηκε. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχίσουμε πίεση, δεν ξέρω, υποστήριξη ε, και στην κυρία Άστον και στον κύριο Φίλε και να πούμε, να διατρανώσουμε ότι και για την ευρωπαϊκή προοπτική ε, αυτό που επιβάλλεται είναι αναθεώρηση του συντάγματος. Τι θα πει η λυπή, the others, θα δώσουμε δηλαδή μια ποσόστοση και για τους άλλους, ένα τέταρτο εκπρόσωπο εκτός από τους τρεις που υπάρχουν ήδη παντού, σε όλα τα πόστα, σε όλους τους οργανισμούς. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ε, χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος οπωσδήποτε. Κάτι άλλο που θα με ενδιαφέρει είναι πώς απαντά ο κύριος Κούκαν ε, σε αυτό που ρώτησε η κυρία Μποσκούρτ, γιατί και ρω... ε, έμαθα και εγώ για αυτό το κόμμα, άκουσα και θέλω να ρωτήσω, έχει τίποτα πιθανότητες στις εκλογές. Ευχαριστώ ο κύριος Κούκαν για να απαντήσει. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για όσα είπατε. Συμφωνώ με όσα είπε η κυρία Πακ αλλά και Λούνατσεκ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η συνέχιση του διαλόγου και πρέπει να είμαστε πιο στεναρή με την καινούργια κυβέρνηση μετά τις εκλογές γιατί σταθερά δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των οποίων και η Βοσνία ρεγοβινη είναι αυτό που απαιτείται για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε κάποια υπομονή, όχι υπερβολική αλλά κάποια για να διατηρηθεί ο διάλογος. Όσο για αυτά που είπε η Χριστίνα Ούλεντς για τον Ντέιτον, καλό θα ήταν να τα σκεφτούμε σοβαρά. Μερικοί πολιτικοί και οι μήκοι ομικρών ε, είπαν ότι η διεθνής κοινότητα ενδυνάμωσε μεν τη συμφωνία, στήριξε τη συμφωνία του Ντέιτον στην αρχή. Αλλά τώρα που υπάρχουν εσωτερικές εξελίξεις δεν είναι εύκολο η διεθνής κοινότητα να τις επηρεάσει. Πράγματι έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε που είχε υπογραφεί η συμφωνία του Ντέιτον και πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο μέλλον Όσο για τις περί, τους περίφημους όρους 5 συν 2 δεν ξέρω πότε θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Αυτά που είπε η κυρία Μποσκούρτ τώρα για το καινούργιο κόμμα Νάσα Στράνκα δεν τους συναντήσαμε όσο δε για το μέλλον τους ε, δεν είμαι και προφήτης, πολιτικός είμαι αλλά θα έλεγα ότι μέχρι τώρα τίποτα δεν δείχνει ότι μπορούν και αυτοί να αλλάξουν, να έχουν κάποια σοβαρή επίπτωση στα εσωτερικά της χώρας. Θα το δούμε, θα φανεί. Αυτά. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και ξανά ευχαριστώ τους συναδέλφους και τα συναδελφάς καθώς και τα άλλα μέλη της ε, αποστολής. Ευχαριστώ. Η κυρία Πάκ ξαναζήτησε το λόγο. Ναι. Εγώ είμαι η συγγήτρια για τη Βοσνία και νομίζω ότι πρέπει να ξαναπάρω το λόγο. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα είναι το εξή. Το Dayton αποτέλεσε τη βάση του νέου κράτους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το Dayton μπορεί να αλλάξει. Όχι εμεί να τα αλλάξουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι δουλειά και ε, αποστολή και καθήκον των κομμάτων και των ε, μερών στην ε, περιφέρεια. Κανένα δεν θα τους εμποδίσει να κάνουν το κράτος τους κυβερνήσιμο εντό εισαγωγικών. Ε, τον ήταν η μόνη λύση να τελειώσει ο πόλεμος. Τώρα έχουν νιωστή φορά εκλογές, μπορούν να τα αλλάξουν, δεν θέλουν να τα αλλάξουν οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να κυβερνηθούν. Ε, θα πρέπει να λάβουν αυτή την πρωτοβουλία. Και εμεί είπαμε, ο ύπατο εκπρόσωπο εκεί, ε, η διεθνή κοινότητα να φύγει, εν περιπτώσει, να μην διοικεί. Αλλά η προπόθεση ακόμα γι' αυτό δεν είναι δεδομένη. Να πω στους συναδέλφους, αλλιώς δεν θα υπάρχει κοινό ε, διαβατήριο. Χαρακτηριστικό για τα αυτοκίνητα, δεν θα υπήρχε σημαία όλα αυτά χωρίς τον Dayton. Δεν θα υπήρχε κοινός υπουργός ε, αμήνης, αν δεν είχαμε αυτή την ε, εκπροσώπηση της διεθνούς κοινότητας, οι ίδιοι πολιτικοί δεν τα κατάφεραν να συνεννοηθούν. Γι' αυτό έχει νόημα ο ύπατος εκπρόσωπος και αυτός να φύγει θέλει, μην νομίζετε. Και ε, θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να φύγει το συντομότερο, αλλά αυτό είναι θέμα των πολιτικών εκεί. Υπάρχουν 7 προποθέσει. 5 συν 2 και αν τι πληρώσουν να φύγει ο άνθρωπο, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και ο, ο πρόεδρος της Βουλής ε, που συζητήσαμε μαζί του μας είπε στο θέμα της θεώρησης των διαβατηρίων μας ε, δώσατε ένα πολύ ε, σαφή οδικό χάρτη. Δώστε μας επίσης ένα οδικό χάρτη τι πρέπει να κάνουμε, ένα φύλλο πορείας για να φτιάξουμε το κράτος. Μα είπαμε εδώ έχετε αυτό το, το μπούσουλα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε ή αν δεν θέλετε να ανταποκριθείτε σε αυτό, τι να κάνουμε. Και σας προειδοποιώ, μην αφήσουμε να εννοηθεί ότι είναι ανασφαλής η χώρα. Δεν ισχύει αυτό. Στη Βοσνία είναι μικρότερη εγκληματικότητα ε, από ό,τι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη της Ένωσης. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είχαμε εχθροπραξίες, πολεμικές ε, ε, σειράξει επιχειρήσεις μεταξύ των εθνοτήτων. Είναι καλό όμως ε, που είναι εκεί πέρα η U4, όχι για να προστατεύει τον οποιονδήποτε, αλλά για να δίνει το μήνυμα ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τη Βοσνία. Και δίνει και ένα υπόβαθρο που μας χρειάζεται εκεί. Παρακαλώ να μην συζητάμε για ανασφάλεια. Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει ανασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως αυτή η συζήτηση Γιατί δείχνει πως συζητήσαμε μάλλον αυτό το σημαντικό θέμα, όμως ε, έχουν όλα αυτά αντίκτυπο και σε άλλα θέματα. Βέβαια αυτό το θέμα ότι το Dayton ήταν έγκυρο για να σταματήσει πια ο πόλεμος, αλλά τώρα αποτελεί πλέον ένα είδος εμποδίου για την πρόοδο της χώρας και αυτό θα πρέπει να το δούμε με λίγες αποχρώσεις. Δηλαδή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα σταθερή. Και δεν θέλουμε προσπαθώντας να κάνουμε το καλό να τα θαλασσώσουμε. Γι' αυτό και προτείνω ο κύριος ε, Κούγκα μου, μαζί με την κυρία Πάκ και αυτός και με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ραμπερτίνη, ε, να ε, συγκεντρώσετε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και να τις απευθύνετε στον ΙΠΑ, το εκπρόσωπο, αλλά και στον Επίτροπο για να είναι πλήρως ενήμεροι και να δούνε επίσης ώρες πώς θα προχωρήσουν. Φαντάζομαι πώς συμφωνείτε με αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ και προχωράμε στο επόμενο σημείο. Και θα ζητήσουμε από τον Λάμσδορφ να παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση είναι για πρώτη φορά στη νέα θητεία, στην 7η Σύνοδο, να πω δύο λόγια. Έχουμε μια ομάδα εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη, όπου συνεργάζονται και συνάδελφοι από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την Επιτροπή Ανάπτυξης, από την Επιτροπή Προπολογισμών κτλ κάνουμε την έκθεση αυτή για να τη δώσουμε στο Συμβούλιο και από τεχνικής πλευράς είναι και σύσταση στο Συμβούλιο για τις προτεραιότητες ε, της Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη για την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα ε, γίνει το φθινόπωρο. Έχουμε άτυπο διάλογο ξεκινήσει ήδη ε, με το αντίστοιχο όργανο του Συμβουλίου, την Ομάδα Εργασίας και χαίρο που με κάλεσαν και εμένα ξανά ως πρόεδρο της δικής μας ομάδας να συμμετέχω στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και να τους παρουσιάσω τα δικά μας συμπεράσματα. Οι πρώτες προτάσεις έχουν μπει ήδη ε, ε, λίγη αύριο το βράδυ, αύριο στις 6 το απόγευμα η προθεσμία για τις τροπολογίες. Έξι είναι τα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι λίγο πιο εκτενές σήμερα, ε, αυτή τη φορά μάλλον, γιατί μετά τη θέση ισχύ ε, της Λισαβόνας αλλάζει η κατάσταση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα, Ευρω... στα Ηνωμένα Έθνη. Τα άλλα θέματα ε, αφορούν την παγκόσμια διακυβέρνηση και μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ειρήνη και ασφάλεια, σας διαβάζω τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στα Ηνωμένα Έθνη. Τι σημαίνει αυτό. Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη πλέον μετά τη θέση σε ισχύ και την κατάργηση της ε, περιτροπής Προεδρίας. Μέχρι τώρα συντόνιζε ένα κράτος μέλος τη στάση μας στον ΟΗΕ. Ε, τώρα έχουμε μία αντιπροσωπεία η οποία δεν έχει ακόμα στελαχωθεί βέβαια, το κάνει τα γραφεία της και ζητούμε ε, να λυθεί αυτό το θέμα στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Το ίδιο ισχύει για διορισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Θέλουμε μεγαλύτερη συνοχή των κρατών μελών και από την αρχή να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Ε, τα επόμενα δύο έτη είναι σημαντικά για τα Ηνωμένα Έθνη. Φέτος θα ε, ελεγχθεί και πάλι το θέμα της, στόχο στόχων της χιλιετίας και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ε, του χρόνου θα αναθεωρηθεί η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εδραίωση της ειρήνης το 2011. Και όποιος γνωρίζει ε, τα Ηνωμένα Έθνη καταλαβαίνει ότι από φέτος αρχίζει η προετοιμασία. Τώρα, η παγκόσμια διακυβέρνηση, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, συνεργάζεται το G20 και ο ΙΕ ίδιος να υπάρχει μια σαφής ε, σύνδεση. Για... Καλό και χρήσιμο το G20, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει ε, στην νομιμότητα και στην παρουσία των ΟΗΕ. Ζητούμε ε, επιτέλους να έχουμε μια συνεκτική πλέον αντιμετώπιση και θέση για το Συμβούλιο Ασφαλείας γίνονται διάφορες προτάσεις για το πώς θα λειτουργήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι προτείνουν διάφορα πράγματα. Η Ένωση είναι βαθιά διχασμένη όπως όλοι γνωρίζουν. Επίσης ε, είναι και το θέμα της αντιμετώπισης του φύλου, ισόρροπης εκπροσώπησης δηλαδή. Ερχόμαστε στο άλλο κεφάλαιο, ειρήνη και ασφάλεια. Ε, βελτίωση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ και συνεννόηση περί την πρόκειται ιδιαίτερα αποστολές θα πρέπει από κοινού να αναλαμβάνουμε μια προσπάθεια, να βελτιώνουμε τη συνεργασία μας και επίσης γνωρίζουμε ότι το DPKO που είναι στη Γενική Γραμματεία επιφορτισμένο με αυτό το θέμα έχει πολλές αποστολές και θα πρέπει να ασχοληθούν και τα κράτη-μέλη με την κατάσταση αυτή. Υπάρχει μια επιτροπή για τη ειρήνευση, Peace Building Commission. Είναι ε, για μένα επιτυχής, θα πρέπει να την ενισχύσουμε και στο ρόλο της και απέναντι ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έρχομαι στο κεφάλαιο της ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αδέλφους εδώ από την Επιτροπή Ανάπτυξης που τα τελευταία χρόνια ε, διαδραμάτισαν πολύ επικοδομητικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μια διάσκεψη για τους στόχους της χιλιετίας θα θυμούν τη συνάδελφοι που είχαμε πάει στη Νέα Υόρκη. Πώς πάμε κάθε χρόνο. Ε, ποιος είναι ο σημαντικότερος στόχος της χιλιετίας όταν ρωτήσαμε. Βέβαια δεν έπεσε κανένα στην παγίδα να πει ότι α, αυτός είναι ο υπαριθμόν ένα στόχος. Αλλά όποιο διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές καταλαβαίνει ότι ο στόχος υπαριθμών 5 που είναι η λεγόμενη μητρική υγεία, δηλαδή η υγεία των γυναικών που αποκτούν παιδιά, είναι πολύ σημαντικός στόχος για τις χιλιετίες. Ε, και γι' αυτό το αναφέρω και εδώ Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ μας βοήθησε και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ένα σημαντικό στοιχείο είναι οι σχέσεις της τρίτης επιτροπής του ΟΗΕ που ασχολείται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το νέο σχετικά συμβούλιο στη Γενέβη που έχει μεγάλες δυσκολίες η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχει μια δυστοκία εκεί η συνεργασία. Και θα πρέπει η τρίτη αυτή επιτροπή να έχει πολύ καλή εκπροσώπηση, καθολική εκπροσώπηση και Για τα ανθρώπινα δικαιώματα αγωνιζόμαστε βεβαίως ε, και στο μέλλον να καταργηθεί η θανατική ποινή, να χειραφετηθούν οι γυναίκες, να ενισχυθούν οι γυναίκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να ενημέρωσω τους συναδέλφους που μπορεί να μην έχουν μάθει ακόμα ότι η νέα ε, ειδική εκπρόσωπος ε, του Γενικού Γραμματέα είναι η πρώην Επίτροπος Μάρκοτ Βάλστρομ. Και για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κτλ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογη, εξαιρετική. Την προωθήσαμε πάρα πολύ την υποψηφιότητά της και χαιρόμαστε που ο, ο, Γενικός Γραμματέας Μπαν Κιμούν ανέθεσε τη θέση αυτή στην κυρία Βάλστρομ. Αλλαγή του κλίματος. Ε, Περιμένουμε ανυπομονησία να δω τι θα γίνει το Μεξικό στο, Δεκέμβριο, στο Μεξικό το Δεκέμβριο, στην COP16. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Γιώ Λάιν, που είναι και πρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντος, ο οποίο πρότεινε να συζητήσουμε κατά πόσο ένα παγκόσμιο φόρουμ μπορεί να έχει αποτελέσματα, Όπω ε, μια τέτοια τεράστια διάσκεψη. εμεί θέλουμε να γίνει στα Ηνωμένα Έθνη ε, αυτό. Αφετέρου είδαμε στην Κοπενχάγη ότι υπήρχαν σφάλματα και οργανωτικά και διαρθωτικά. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον και τα κράτη-μέλη που σύμφωνα με το χάρτη των ε, Ηνωμένων Εθνών και το άρθρο 2 είναι μέλη αυτής της παγκόσμιας ε, οργάνωσης. Αυτά εν συντομία ως συστάσεις προς το Συμβούλιο. Σας είπα προθεσμία κατάθεση τροπολογιών λίγη αύριο στις 6 το απόγευμα. Αν έχετε ρωτήσει σχόλια με χαρά να τα απαντήσω. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Λάμστον για το έργο του και στη Νέα Υόρκη και για την έκθεση. Είναι πάρα πολύ καλή η σύνθεση που έχει κάνει στο σχέδιο έκθεσης του γιατί είναι πολύ μεγάλο το φάσμα, η βεντάλια των θεμάτων που διαπραγματεύεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και... Και ο κύριος Λάμστροφ ε, πραγματικά συνεργάστηκε πολύ καλά, πολύ ικανοποιητικά με τις πολιτικές ομάδες και μάλιστα έχει συμπεριβάλει και δικά μας συμπεριλάβει ε, σχόλια. Ωστόσο, εγώ θα κάνω και κάποιες τροπολογίες και το ανακοινώνω ήδη εδώ μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στην ενιαία ε, φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ απαραίτητη ε, μετά τη συνήθιση της Αβώνας να ακούγεται η Ένωση με μία φωνή και επειδή έχουμε και εμπειρίες και διδάγματα από τη διάσκεψη Κοπεχάγης για την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να τα καταγράψω αυτά σε κάποιες τροπολογίες για τους όχους άλλα Άλλοι στόχοι είναι πιο ευρύς, ενώ οι στόχοι της χιλιετίας όμως είναι συνολικό πακέτο, δεν μπορούμε να τους διαχωρίσουμε. Και σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική θα πρέπει να ενισχύσουμε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στη θεσμική μεταρρύθμιση του οργανισμού. Επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη προβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της δεκάτης επαιτίου ε, του ψηφίσματος 1325 για την ισότητα των φύλων. Αυτά. Κατά τα άλλα, οι συστάσεις και έκθεση του κυρίου Λάνστροφ είναι πάρα πολύ πλήρης και συμπεριλαμβάνει και τις ανησυχίες και τα μελήματα των άλλων πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίλαν και Μόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Κόμι Λάμστορφ για το κείμενό του. Είναι πολύ πλήρες, είναι πολύ ισόρροπο και χαίρομαι που έχει συμπεριλάβει και ε, προτάσεις δικές μας στο αρχικό κείμενο που κυκλοφόρησε στις 8 Φεβρουαρίου. Στο Στρασβούργο είχαμε συνεδριάσει και κάναμε κάποιες προτάσεις τις οποίες έλαβε υπόψη ο εισηγητής. Προσωπικά θα κάνω και εγώ μερικές μικρές τροπολογίες που δεν επηρεάζουν την ουσία της έκθεσης. Τη μία την ανέφερε ο κύριος Λάμστορφ, η ανάγκη να πούμε ποιοι είναι οι πυλώνες ε, του ΟΗΕ στο τμήμα Β ε, και ποια, ποιοι είναι οι στόχοι. Η ειρήνη, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Επίσης, θα αναφερθώ στην Παγκόσμια Σύμβαση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βέβαια, ήδη έχει κάποιες αναφορές στο κείμενο, αλλά νομίζω ε, καλό θα ήταν να αναφέρεται πιο ρητά για να είναι πλήρης. Και θα κάνω και μια τροπολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Λάμστροφ, για το πληρέστατο κείμενο και την ισόρροπη προσέγγιση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνετε, να κάνετε. Η κυρία Λόκμπιλερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Είναι πολύ καλή έκθεση. Μία συμπλήρωση θα ήθελα να προτείνω εγώ μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν αλλά και στο παρόν ε, εργάζεται πάρα πολύ διεθνώς για την κατάργηση της θενατική ποινής. Και ε, είναι και επιτυχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υποχωρεί η θενατική ποινή παγκοσμίω. Ξέρουμε ότι παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε τρομακτικές καταστάσεις, αλλά δεν θα πρέπει ε, απλώς να τα παριθμούμε αυτά, να πούμε καταπολέμηση και κατάργηση των βασανιστήριων. Γιατί, Γιατί το βασανιστήριο πραγματικά παραβιάζει, βιάζει την προσωπικότητα του καθενός και είναι σε κατάφορη αντίφαση με τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα του κάθε του κάθε προσώπου ξεχωριστά, του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να συμπεριλάβετε και την πρόταση που λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παντού, γενικώ ε, στη Γενική Συνέλευση των Μένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καταπολέμηση των βασανιστήριων. Φέτος είναι και επίκαιρο γιατί ο ειδικό εισηγητής ε, Μάνφρετ Νόβακ κατά ε, των βασανιστήριων ολοκληρώνει την επιτυχή του πενταετή θητεία και θα ήταν σημαντικό να στείλει ένα μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μας ενδιαφέρει πολύ κατά πολέμηση των βασανιστήριων και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί μεταξύ άλλων, μας ενδιαφέρει Σε Ευχαριστώ. Κύριος Μαύρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λάμσντορφ, τον οποίον και συγχαίρω, αλλά θα κάνω μια πετροπολογία στο κείμενο. Στο σημείο που αφορά τις συστάσεις που απευθύνουμε Πολύ συγκεκριμένο το σημείο που θεωρώ πως δεν ε, καταφέρνουμε να κάνουμε πραγματικά προτάσεις. Είναι εκείνο το κομμάτι του κειμένου που αφορά την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλής. Γιατί το να λέμε, όπω λέει στο κείμενο, ότι παραμένει ένα ε, μακροπρόθεσμος στόχο, η λέξη μακροπρόθεσμος ε, μοιάζει πολύ με τη λέξη ποτέ. Ε, οπότε το να επαναλαμβάνουμε αργότερα ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί χωρίς να ζημιωθεί το κύρος και το βάρος των κρατών μελών στο εσωτερικό αυτού του οργάνου δεν καταλαβαίνουμε αν παραμένει ίδιος, αν παραμένει ο ίδιος ο ρόλος των κρατών μελών ε, τι νόημα έχει να έχει έδρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άρα λοιπόν εγώ θα προτείνω να καταργηθούν, να διαγραφούν αυτά τα κομμάτια τα οποία σας ανέφερα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Κύριε Λάμσντορφ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια των συναδέλφων. Με χαρά και με ενδιαφέρον περιμένω τις τροπολογίες. Ορισμένα θέματα ήδη τα ε, εγκρίνω νοερός, ειδικά αυτά που είπε η κυρία Λόχμπίλερ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι Αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριο Μάουρο τώρα. Τι να σα πω. Ναι, με ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο κάπου να διαμορφώσει θέση για το θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάμε για την αναθεώρηση των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε πλήρως την καρδιά την ίδια των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνάδελφοι που εργάστηκαν σε αυτό το θέμα και από την περασμένη θητεία όπως ο συνάδελφος Μιγιάν Μπον και άλλοι θα γνωρίζουν ότι στο παρελθόν λέγαμε πολύ ε, πιο λεπτομερή πράγματα, πιο σημαντικά και μάλιστα ε, είχαμε και διαπληκτιστεί για το μοντέλο. Γιατί ε, θέλουμε ε, ως χώρες, γιατί δεν θέλουμε το ίδιο πράγμα ως χώρες και γι' αυτό διαπληκτιστήκαμε πολύ. Τώρα, συνειδητά μετά τη θέση σε ισχύ της Λισαβόνας, κάνουμε και πάλι μια έκκληση στα κράτη-μέλη και στην ύπατη εκπρόσωπο να καθίσουν σοβαρά και να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια κοινή θέση, εν περιπτώσει, για το θέμα αυτό, για να ε, πάμε στη Γενική Συνέλευση ενωμένη. Δεν είναι καλό να μην μπει τίποτα το κοινοβούλιο απολύτω να το αποσιωπήσει, να καλέσει τα κράτη-μέλη. Έτσι κι αλλιώ το όλο κείμενο είναι μια σύσταση στα κράτη-μέλη. Να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το θέμα και να κάνουμε μια προσπάθεια σοβαρή όμω να καταλήξουμε σε κοινή θέση για το Συμβόλιο Ασφαλεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα βρει σύμφωνο, αν όχι όλου του συναδέλφου, την πλειοψηφία του. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με μεγάλη συνένεση και θα μπορέσουμε να τα ψηφίσουμε και στο τέλος. Ευχαριστώ. Very much. So... Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών αύριο στις 6 το απόγευμα. Ωραία λοιπόν, προχωράμε και έχουμε και μια έκθεση της κυρίας Λόχμπιλερ για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τι εκβιομηχανισμένε χώρες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ζητήθηκε την περασμένη φορά να συντάξω ένα σχέδιο χνομοδότησης και έκτοτε είχαμε μία συνεδρίαση με την Κομισιόν για να συζητήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες αυτό το σχέδιο. Κάναμε και μία δεύτερη συνάντηση με τους σκιώδεις ηγητές της ΑΦΕΤ. Για τα περισσότερα θέματα που συζητήσαμε και θίξαμε, ε, συμφωνούσαμε για μια νέα διατύπωση ή για τις συγκεκριμένες προτάσεις. Οπότε τώρα έχουμε ενώπιόν μας ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, 8 τον αριθμό, και ε, που βασικά προέρχονται από μένα που είμαι η συντάκτρια και δείχνουν τη συνένεση στην οποία καταλήξαμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει άλλες γραπτές τροπολογίες και εν συντομία θα ήθελα να σας τις ε, περιγράψω. Έχουμε λοιπόν την τροπολογία 21 όπου προσθέτουμε μόνο ποια είναι η νομική βάση. Έχουμε επίσης την τροπολογία 22 όπου αναφέρεται το θέμα του νέου ονόματος του μέσου, πράγμα που επίσης συζητήσαμε τελευταία φορά στην ΑΦΕΤ. Και να υπογραμμίσω ότι το όνομα βέβαια δεν είναι το πιο σημαντικό θέμα, αλλά είναι καλύτερο να έχει ένα νέο τίτλο ώστε να καλύπτεται ο ευρύτερος, το ευρύτερο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και γι' αυτό αποφασίσαμε να καλείται μέσω συνεργασίας με χώρες στη Μέση Ανατολή, Ασία, Αμερική και Νότια Αφρική. Να σα πω από αυτού ότι ο εισηγητής τη ΣΥΝΤΑ δεν συμφωνεί με την ονομασία αυτή. Τώρα, στην ε, τροπολογία 23... Ε, υπάρχει ένα μικρό λάθος που λέει ότι ο νέος κανονισμός θα πρέπει να στηρίζει την οικονομική συνεργασία αντί την ε, κοινωνικο-οικονομική συνεργασία και έχουμε προσθέσει και την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και της πανεπιστημιακής συνεργασίας. Εξίσου σημαντικό είναι να πούμε ότι η τροπολογία θα πρέπει να κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο Μηχανισμό Αναπτυξιακή Συνεργασία DCA και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια το νέο μέσο που θα καλύπτει ε, ε, ε, συμφέροντα αναπτυξιακά και δεν θα είναι στο ODA. Στην ε, τροπολογία 24 μιλάμε για συνεργασία με εταίρους ε, που έχουν παρόμοιες ε, πολιτικές, οικονομικές δομές αλλά και αξίες. Αν δούμε την ομάδα των χωρών που εμπίπτουν σε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας θα πρέπει σαφώς να πούμε πως δεν έχουμε παρόμοιες δομές και πως πολλές φορές δεν προωθούν ε, τις ίδιες αξίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνήσαμε λοιπόν με την Κομισιόν να κάνουμε μια καλύτερη περιγραφή και λέει λοιπόν η συνεργασία αποσκοπεί σε σύμπραξη με χώρες εταίρους προς επίτευξη των εξής στόχων. Άμβληση της σύγκρουσης και τόνος του διαλόγου και προσέγγισης, ημερισμός προμπαρομείων ε, πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών δομών και αξιών και προαγωγή αυτών, και ε, αύξηση των ανταλλαγών με σημαντικούς ε, τέρους και παράγοντες σε διμερή βάση, σε πολυμερή φόρα και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Και επίση θα πρέπει να πω πω από αυτό το σημείο η ΙΝΤΑ έχει διαφορετική άποψη γιατί θα ήθελε να συνεργαστεί και να το έχει αυτό ε, υπό όρου. Στην τροπολογία 25 προσθέτουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα διευρυμένο ε, πεδίο εφαρμογή ε, τίου μέσου ε, με έμφαση στις δραστηριότητες προς αποσόβηση της αλλαγής του κλίματος και τα πυροβολοντικά και κοινωνικά βιώσιμες καθαρές και προσαρμοσμένες τεχνολογίες. 26 λέμε για την ε, παρότρινση της οικονομικής συνεργασίας και με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έπειτα στην τροπολογία 27 περιγράφουμε πιο συγκεκριμένα την πρόθεση των ε, ε, συνεταιριστικών σχεδίων των σχεδίων μάλλον συνεργασίας στον τομέα ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, να σας πω ότι εμείς εδώ στην τελευταία τροπολογία επιμένουμε στο αρχικό κείμενο και υπογραμμίζουμε ότι υπάρχει διάκριση στον προπολογισμό από το 2007 μέχρι το 2013 που σχετίζεται ήδη, με ήδη λιμένες αποφάσεις αλλά είναι επίσης απαραίτητο να τονίσουμε ότι από το 2013 και μετά θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε και ίσως να βρούμε και άλλες λύσεις. Έχουμε μία διαφωνία με τον γιατί ο κύριο Γκάλερ από την ΑΦΕΤ, διότι Υποστηρίζουμε τη θέση πως η χρηματοδότηση ε, δεν θα πρέπει να μεταφερθεί από το μέσο DCI. Τέλος, να συστήσω ότι η ΑΦΕΤ θα αναζητήσει την υποστήριξη και της Λέδης ε, Άστον για το πώς αυτό το μέσο το οποίο φτιάχνει τα θεμέλια για ένα μελλοντικό μέσο για την εξωτερική πολιτική, πώς θα είναι αυτό το μέσο μετά αυτή την ενδιάμεση περίοδο, δηλαδή από το 2013 και μετά, όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά και τον προϋπολογισμό του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος πως η διαβούλευση θα είναι ιδιαίτερα καρποφόρα και τις δύο πλευρές και ζητώ τώρα από τον κύριο Γκάλε να πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά τη συνάδελφο Λόχ Μπίλερ. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνεργασία και θέλω και την Κομισιόν να την ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια συνάντηση πολύ καρποφόρα. Και πρόθεσε και τη συνένεση και στους δύο τομείς. Το είπε και η συνάδελφος ήδη. Υπάρχει ένα σημείο που διαφωνούμε. Για τους επιπλέον πόρους για τις νέες ε, αποστολές. Εμείς έχουμε τη ρητή άποψη που λέει όταν περνάει ένα πεδίο ε, καθηκόντων υποχρεώσεων από το ένα κεφάλαιο, από το ένα μέσο στο άλλο, θα πρέπει κάπου να βρεθούν και τα λεφτά. Δηλαδή τα χρήματα ακολουθούν ε, τις υποχρεώσεις. Αν δεν απατώμε, είναι η τροπολογία 28 αυτή. Αυτή δεν θα την υπερψηφίσουμε, δεν μπορούμε. Αλλά κατά τα άλλα συμφωνούμε πολύ. Και αν η Επιτροπή έρθει στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια και κάνει μια εξήγηση για τη διαφύλιξη των ε, συμφερόντων και των ενδιαφερόντων μας ως προς την επιτροπολογία, μπορεί να αποσύρουμε και καμιά τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you. Now, um, Mr. Panzeri, please. Panzeri. Grazie, Presidente. Devo dire molto brevemente che a nome dei socialisti e dei democratici... Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρέπει να πω στο όνομα των ε, να προφανώς ευχαριστώ την, ε, την ε, εισηγήτρια για την εργασία που έκανε. Νομίζω πως οι επαφές που είχαμε έφεραν ένα, κατέληξαν σε ένα θετικό μάλλον αποτέλεσμα και η ικανότητα της εισηγήτριας να εισακούσει τις επιθυμίες μας ε, βοήθησε βέβαια σε αυτό και αυτό και εμείς συμφωνούμε με όλα τα σημεία τα οποία σας παρουσίασε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μουνιέ από τη Γενική Διεύθυνση Ρελέξ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για τον διάλογο που είχαμε μαζί του και οι περισσότερες τροπολογίες θα γίνουν δεκτές από την Κομισιόν αφού βέβαια τις εξετάσει αλλά γενικά δεν θα υπάρξει νομίζω πρόβλημα. Βέβαια υπάρχει ακόμη το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εμείς θεωρούμε ότι οι ετήσιες διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού μπορούν να το λύσουν και οι πληρωμές δεν χρειάζεται να μπουν ήδη στο σώμα του νομοθετικού, της νομοθετικής πράξης, μπορεί να βρεθεί μια λύση άλλη. Όσο για τις τροπολογίες τις υπόλοιπες, Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει τις επόμενες εβδομάδες και πρέπει και αυτό κάποτε κάπως να λυθεί. Χρειάζεται βέβαια μία άμεση προσαρμογή του εργαλείου αυτού για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και όσες δραστηριότητες έχουν ήδη αναλυφθεί και εφαρμόζονται πρέπει φυσικά να μπορέσουν να συνεχιστούν. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια συμφωνία σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λότμπίλερ. Ε, και εγώ ευχαριστώ για την επικοδομητική μας συνεργασία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Θα φανεί και από την ψηφοφορία το απόγευμα. Ευχαριστώ. Κι εγώ, κι εγώ. Καιρός είναι τώρα να περάσουμε στο θέμα του κυρίου Κόβαλ που ήταν πρόεδρος της αντιπροσωπείας παρατήρησης των εκλογών στην Ουκαρανία. Έχει το λόγο. Yes, yes. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν επικεφαλής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιτήρησης των Εκλογών στην Ουκρανία. Και κατά τους δύο γύρους επισκεφθήκαμε πολλά εκλογικά τμήματα και στο Κίεβο και στο Ντονιέτσκο. και τα συμπεράσματά μας εμφαίνονται στην αναφορά που υποβάλαμε. Ιδίως σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές στην Ουκρανία, η αποτίμησή μας ήταν θετική και νομίζω ότι οι εκλογές αυτές πρέπει πάρματι να θεωρηθούν ως καλύτερες από εκείνες που έγιναν σε πολλές πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Οι προηγούμενες επίσης είχαν αποτιμηθεί θετικά, αλλά η Ουκρανία είναι από τις λίγες χώρες της Σοβιετικής περίοδου που έχουν οργανώσει εκλογές με παρατηρητές. Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα διότι η Πολωνία ακόμη δεν έχει αποδηθεί της παλαιάς, της, των παλαιών της συνηθιών της, του ολοκληρωτισμού. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε βέβαια ούτε τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν, οι κυριότεροι από τις οποίες ήταν η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ουκρανία. Και η ίδια η εκλογική διαδικασία βέβαια είχε μερικές ελλείψεις. Από συζητήσεις, με συζητήσεις πρέπει να συνεχίσουμε και επαφές να το τονίζουμε γιατί η, τα εκλογικά πρότυπα, οι εκλογικές διαδικασίες είναι κάτι που πρέπει να λειτουργήσει απρόσκοπτα κυρίως με καλύτερη χρηματοδότηση της πολιτικής ζωής στην Ουκρανία. Γιατί χωρίς αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει πρόοδος ούτε σε επόμενες εκλογές. Επίσης πρέπει να τονίσουμε και ορισμένα ελάσσονα θέματα που όμως ενδιέφεραν πολύ το κοινό παραδείγματος χάρη τις προσαρμογές της του εκλογικού νόμου σύμφωνα με την Διεθνή Ομάδα Παρατήρησης οι ελλείψεις που σημειώθηκαν δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα σημαντικά αλλά επηρέασαν το κλίμα της προεκλογικής περίοδου η ψηλή προσέλευση και στους δύο γύρους είναι επίσης αξιοσημείωτη. Οι διάφορες αποτιμήσεις που έγιναν δεν το τόνισαν αυτό ιδιαίτερα γιατί παρόλα αυτά αυτό διαφοροποιεί την Ουκρανία από πολλές εκλογές και σε ενωσιακές ακόμη χώρες. Οι Ουκρανοί γενικά έχουν εμπιστοσύνη στην διαεκλογική διαδικασία. Αυτό φαίνεται. Και βέβαια αυτό συνδυάζεται με την αποτελεσματική και αξιοπρεπή διαδοχή στην εξουσία που έγινε με ομαλότερο τρόπο από ό,τι οι άλλες πρώην Σοβιετικές χώρες. Λόγω της υψηλής προσέλευσης δε, φαίνεται ότι ο κόσμος παίρνει πολύ στα σοβαρά και η πολιτική την πολιτική ζωή. Και άρα πρέπει να δηλώσουμε ότι η Ουκρανία είναι πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα που αν που υπό ορισμένου όρους θα μπορούσε να έχει και ευρωπαϊκή προοπτική, όχι στο άμεσο μέλλον βέβαια, αλλά πάντως το καλύτερο στοιχείο που έχουμε να τονίσουμε είναι η υψηλή εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις εκλογές. Αυτό πρέπει να φαίνεται και στις συμφωνίες που θα συνάψουμε με την Ουκρανία. Γιατί οι πολίτες έχουν κάνει προσπάθειες και πρέπει να βραβευθούν η κοινωνία των πολιτών ε, παίζει σημαντικό ρόλο και οι δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να τους πούμε ότι μπορεί τελικά να καταλήξουν και σε συμμετοχή στην Ένωση. Εμείς οι κοινοβουλευτικοί πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να απελευθερώσουμε το καθεστώς των θεωρήσεων, ίσως και να τις καταργήσουμε. Τώρα, το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών παραμένει. Η δική μας ανταπόκριση στην υψηλή προσέλευση θα έπρεπε να είναι η δήλωση ότι πρέπει να διευκολυνθεί το καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα βέβαια όπως οι επαφές μας γενικότερα με την Ουκρανική κοινωνία. Και τέλος θέλω να τονίσω τον ρόλο που έπαιξαν οι διάφορες παρατηρητικές αποστολές κατά τις εκλογές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο μόνος θεσμός που είναι πάντοτε παρόν σε τέτοιες περιστάσεις. Επίσης πρέπει να τονίσουμε το ρόλο άλλων οργανώσεων που βοήθησαν και μας. Γιατί θα ήταν απαραίτητο γιατί έτσι φαίνεται μπορούμε να πούμε ότι παρακολουθήσαμε όλες τις πτυχές της εκλογικής διαδικασίας. Και ευχαριστούμε τον πρέσβη Γκαντζοβίν, που έκανε τόσα πολλά για να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα. πρέπει να γίνουν νομίζω συνομιλίες μεταξύ όλων των αντιπροσωπιών που παρατήρησαν εκεί τις εκλογές μεταξύ των οποίων και το ΝΑΤΟ για την ενδυνάμωση της μελλοντική συνεργασίας για τέτοιες αποστολές. Εγώ δεν ήθελα οι εκπρόσωποι της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών να συμμετέχουν με ίσους όρους με τη δική μας αντιπροσωπεία, αλλά δεν αποκλείει αυτό μια συνεργασία με τους εκπροσώπους αυτούς. Χρειάζεται συνεργασία, είναι απαραίτητη. Και τέλος, Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες, ιδιαίτερα τον Στέφαν Βίτσνερ και την ομάδα των υπευθύνων ασφαλείας. Όλοι αυτοί συνέβαλαν στην επιτυχία της αποστολής έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είχε κάποια αξία. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της αποστολής αυτής. Είναι πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο να επιτηρεί τέτοιου είδου εκλογές. Στην Ουκρανία η αποστολή θεωρήθηκε πολύ σημαντική και, για τους δύο, και κατά τους δύο γύρους. Πριν φτάσουμε πριν πάμε στην Ουκρανία, είχε παρατηρηθεί κάποια πόλωση, κάποια ένταση. Και το ίδιο και πριν από το δεύτερο γύρο. Αλλά κατά την ίδια την ημέρα των εκλογών παρατηρήσαμε πολύ βελτιωμένο κλίμα και μεγάλη πρόοδο και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τα συμπεράσματά μας και άλλων παρατηρητικών αποστολών είναι παρόμοια. Η Όντιρ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και πολύ διαφανή, πολύ διαφανή ρόλο έπαιξε. Όχι ότι ήταν ενιαία όλα τα πρότυπα, αλλά παρόμοια. Οι εκλογές λοιπόν στην Ουκρανία δεν μπορούμε να πούμε ότι μειώνουν την ανάγκη να προσέχουμε τα πράγματα παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, και εγώ, όλοι είναι πεπισμένοι ότι η Ουκρανία είναι σημαντική χώρα και ότι οτιδήποτε συμβεί εκεί επηρεάζει και μας. Άρα πρέπει να προσέχουμε τι συμβαίνει εκεί. Ελπίζουμε και εμείς οι εκλογές αυτές να καταλήξουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα και βελτίωση. Αυτά που είπατε δε είναι σημαντικά. Λοιπόν, Κύριε Κόβαν θέλετε να απαντήσετε ή όχι μήπως. Ε, λίγο, λίγο. Δύο μόνο θέματα, Πρόεδρε, που είχα ξεχάσει να τα αναφέρω προηγουμένως. Ξέχασα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους και βουλευτάς από άλλες πολιτικές ομάδες με τους οποίους είχαμε εξαιρετική συνεργασία και να σας καλέσω στο αυριανό μας σεμινάριο της ΕΠΕΞ με την Ουκρανική Αντιπροσωπεία αύριο στις 10. Εκεί θα μπορέσουμε να ακούσουμε και άλλους εμπειρογνώμονες επί Ουκρανικών θεμάτων. Εκεί νομίζω θα βγουν θετικά συμπεράσματα για όλη μας την αποστολή. Ο δε πρόεδρος Βίκτορ Γιαννούκοβιτς θα αναλάβει τα καθήκοντά του παρουσία πάλι της αντιπροσωπείας μας. Ε, καλό και εγώ όλους τους συναδέλφους αύριο στο σεμινάριο μεταξύ 10 και 12 που θα αναφέρει τα ίδια θέματα. Λοιπόν, τώρα το τελευταίο θέμα του πρωινού η μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκαρανία. Ο κύριος Ρίσαρντ Άντωνι Λεγκούτκο. He was not seated. He has to sit. uh, Thank you, Mr. Chairman. Uh, As a rapporteur, I believe that the Committee on Foreign Affairs. Νομίζω πως ε, η Επιτροπή ΕΦΕΤ θα πρέπει να προωθήσει το θέμα της, μακροοικο... της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία ε, δεδομένου του αντίκτυπου που είχε η κρίση στην χώρα αυτή τον περασμένο χρόνο. 15% μείον στο ΑΕΠ. Πρόκειται για 5 εκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή δανείου που στόχο θα έχουν να συμβάλλουν στις γενικές ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών της Ουκρανίας και τις εξωτερικές ανάγκες χρηματοδότησης του κρατικού προπολογισμού όπως, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να θυμίσω επίσης ε, ότι 110 εκατομμύρια ευρώ που χορηγούνται από την απόφαση του Συμβουλίου του 2010 2002, ε, συγγνώμη, αλλά αυτή η απόφαση δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Ωστόσο, προτείνω να τροποποιηθεί με οκτώ τροπολογίες το σχέδιο της Επιτροπής με τους εξής στόχους υπόψη. Πρώτος στόχος είναι να βελτιωθεί η συνοχή των Ευρω... της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης. Σε αρκετέ περιπτώσεις η Κομισιόν έχει συντάξει τις πρώτους όρους στους οποίους έχει συμφωνήσει και η Ουκρανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πιστεύω πως οποιαδήποτε βοήθεια κοινοτική που δίνεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να είναι συνεπίση με τις προτεραιότητες των πολιτικών της Ένωσης και της συγκεκριμένης χώρας εταίρου. Γι' αυτό και προτείνω να τροποποιηθεί το κείμενο ώστε αυτό να συμφωνεί με την ατζέντα σύνδεσης της Ένωσης με την Ουκρανία που συμφωνήθηκε το 2009 και καλύπτεται από τις τροπολογίες 1, 3, 5 και 6. Δεύτερος στόχος είναι να αυξηθεί ο ρόλος της Ένωσης ώστε να πυροδοτηθούν οι απαραίτητες διαθετικές αλλαγές, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το ρόλο και τις ε, σημερινές σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Ουκρανίας που συμπεριλαμβάνουν την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση και ε, ε, ολοκλήρωση την, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για τους όρους θα ήθελα να προτείνω την εισαγωγή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, χρονικών πλαισίων μέσα στους όρους. Άρα θα πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι όροι πριν από την ε, απελευθέρωση της βοήθειας. Αυτό καλύπτονται από τις τροπολογίες 6 και 7. Τρίτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, προϋπόθεση εκ των νόνου Κάνεφ ε, απελευθερώνεται οποιαδήποτε βοήθεια, δηλαδή η συνένεση των Ουκρανικής πολιτικής ελίτ ε, να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να συνεχίσει τις ε, μεταρρυθμίσεις. Και σε αυτό αναφέρομαι στην τροπολογία 2. Τέταρτον, τέλος, πιστεύω πως είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά μέσω κατά τη διάρκεια μάλλον της πορείας εφαρμογής και ακόμα περισσότερο γιατί αυτό θα υιοθετηθεί μέσω της ε, κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και αυτά καλύπτονται από τις τροπολογίες 4 και 8. Δύο παρατηρήσεις για το χρονοδιάγραμμα. Δεδομένου ότι η ΙΝΤΑ είναι η επί της αρμόδια επιτροπή και ψηφίζει στις 16 Μαρτίου, θα ήθελα να σας θυμίσω λοιπόν ότι πρέπει να δουλέψουμε εντός ενός πολύ στενού χρονικού περιθωρίου και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται στην 1η Μαρτίου 6 το απόγευμα. Και η ψηφοφορία, όπως είπαμε, γίνεται στις 16 Μαρτίου στην Ίντα. Συνάδελφοι, προσβλέπω στα σχόλιά σας και τις απόψεις σας και ευχαρίστως ε, συνεργαστώ μαζί σας για το θέμα αυτό, αλλά και για τα επόμενα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είτε πολύ γρήγορα πάμε, είτε πολύ ώρα, πολύ αργούμε. Ε, μάλλον σήμερα πήγαμε πολύ γρήγορα και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή δεν είναι εδώ για να σχολιάσουν έκθεση. Είμαι βέβαιο πώ θα υπάρξει επικοινωνία με κάποιο τρόπο. Και αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, τώρα είναι η ώρα. Όχι. Σα ευχαριστώ πολύ. Να πω άλλη μια φορά αυτά που είπε ο εισηγητή, ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η 1η Μαρτίου, 18 η ώρα δηλαδή 6 το απόγευμα και όπως είπατε η ψηφοφορία στην 90 θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Τώρα, απόψε το απόγευμα θα ξεκινήσουμε στις 3 με την ακρόαση για την Ένωση για τη Μεσόγειο και ψηφοφορίες θα γίνουν γύρω στις 4 και 4. Οπότε κανονίστε τα προγράμματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε